για την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, dear Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Η έκθεσή μας προσπαθεί να σπάσει δύο ηλίθια αλλά διαδεδομένα στερεότυπα. Το πρώτο είναι ότι η ψηφιοποίηση αφορά μόνο τις τεχνολογικές εξέλιξεις. Όχι. Η ψηφιοποίηση θα διαμορφώσει εκ νέου τις κοινωνίες μας και θα επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής μας. Οπότε η ψηφιακή πολιτική είναι κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς η ισότητα θα πρέπει να είναι στην καρδιά αυτής της συζήτησης. Το δεύτερο είναι ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για την ψηφιακή επανάσταση. Ενδιαφέρονται λοιπόν, σας το λέω εγώ. Γράφοντα αυτή την έκθεση μίλησα με πάρα πολλέ γυναίκε που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο και εγώ πίστηκα. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια στον τομέα της πληροφορικής ή στην εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις σωστές προϋποθέσεις για να κατακτήσουν πλήρως τον ψηφιακό κόσμο. Τα ηλίθια αυτά στερεότυπα δεν είναι η μοίρα μας. Δεν είναι γραφτό. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό ακριβώς κάνει αυτή η έκθεση επειδή η έκθεση πραγματικά δείχνει ποιες είναι οι προκλήσεις αλλά δίνει και συγκεκριμένα εργαλεία για να τα ξεπεράσουμε και δείχνει τις εκπληκτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τις γυναίκες και την ισότητα στις κοινωνίες μας. Εάν η Βουλγάρα η οποία φτιάχνει παιχνίδια κάθε μέρα καταφέρει να ξεπεράσει μια Γαλλοκαμερουνέζα η οποία κάνει την ίδια δουλειά ή θα μπορούσε παραδείγματο χάρη να βοηθήσει μια Ιρλανδέζα την οποία παρενοχλεί ένα τρόλ στο facebook. Αυτή η έκθεση απαντάει σε όλα. Ζητάει περισσότερη χρηματοδότηση για γυναίκες επιχειρηματίες και ζητάει καλύτερη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών για να καταπολεμηθεί η παρενόχληση στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε βλέπουμε πως τα μέσα υπάρχουν. Τώρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να τα χρησιμοποιήσουμε. Και κυρία Γιούροβα, ελπίζω όχι μόνο εσείς, αλλά ολόκληρη η Επιτροπή να σταθεί στο πλευρό μας και να τα προωθήσει αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που βλέπουμε σε αυτή την έκθεση δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την βοήθεια ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, γυναικών επιχειρηματιών και πολλών άλλων που μας βοήθησαν και τη δουλειά βεβαίως των συναδέλφων που παρακολουθούσαν αυτή την έκθεση, των σχεδόν εισηγητών δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την επικοδομητική εργασία. Νομίζω πως μπορούμε πραγματικά να οικοδομήσουμε μια ουσιακή ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους πάντες και θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες. Και ελπίζω έτσι να έχουμε μια αφετηρία και μια ευρεία πλειοψηφία αύριο. γιατί βεβαίως αύριο είναι και η μέρα των κοριτσιών στην πληροφορική. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Στο Catch the Eye. Η κυρία Κομοδίνη έχει το λόγο. Μια ισχυρή ψηφιακή οικονομία είναι πολύτιμη για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και των γυναικών. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός κυρίως των νέων κοριτσιών έχουν αρχίσει να αναζητούν στα σταδιοδρομία στα ηλεκτρονικά, στην ψηφιακή οικονομία. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ο ψηφιακός τομέας είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στο οικονομικό αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξει σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση και για τις ε, νέες γυναίκες να συμμετέχουν στις εξελίξεις και να κατανοήσουν ότι συμμετέχουν στην ψηφιακή καινοτομία και είναι σε θέση να αποκτήσουν τις ε, δεξιότητες που απαιτούνται και διαμέσου επίσης της διαβίου κατάρτισης θα βοηθηθούν οι γυναίκες να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες απουσιάζει. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή και η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας είναι αναγκαίες όσο ποτέ. Αρχικά στα κράτη-μέλη της Ένωσης παρατηρούμε ότι μόλις το 9% των προγραμματιστών είναι γυναίκες, ενώ μόνο το 19% των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας έχουν γυναίκες διευθύντριες, σε σχέση με το 45% των εργαζομένων σε άλλους τομείς αυτό φυσικά είναι αποτέλεσμα του σημαντικού χάσματος που υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας. βέβαια οι διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων φαίνονται και στον εργασιακό χώρο γενικότερα αφού οι μισθολογικές διαφορές και οι διαφορές στις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλες ενώ σε χώρες όπως η ελλάδα που πλήττεται από τα μνημόνια οι γυναίκες αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού που έχει πληγεί περισσότερο είναι επομένω αναγκαίο να προωθηθεί η ισότητα των δύο φύλων στον τομέα τη ψηφιακή οικονομία να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών σε ηγετικέ θέσει και να εξαλειφθεί κάθε μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην εργασία. ευχαριστώ. Ο κύριος Δυστυχώς ε, και η ψηφιακή εποχή σήμερα ε, περιλαμβάνει ανισότητα ε, σε μια εποχή που η γεωργία θα έπρεπε να είναι σημαντική ή, την βιομηχανική εποχή που είχαμε τις μηχα... μηχανές που μας βοηθούν ε, από τότε είχαμε ε, ανισότητα, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα που έχουμε την ψηφιακή εποχή, που έχουμε την πρόοδο. Είναι σημαντικό λοιπόν να χειραφετήσουμε τις γυναίκες και να έχουμε, εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε ψηφιακό γραμματισμό των κοριτσιών και γυναικών γιατί σήμερα έχουμε πολλά και καλά παραδείγματα. Πολύ ευχαρίστω θα υπερψηφίσω την έκθεση γιατί ε, μιλά για μια και δική μου πεποίθηση, την ανάγκη της πρόσβασης στην ψηφιοποίηση. Θα πρέπει ε, να δώσουμε και να δείξουμε τα θετικά παραδείγματα, τα παραδείγματα προς μίμηση. Ποια είναι τα καλά παραδείγματα, ποιες είναι οι καλές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού επέτυχαν οι γυναίκες και σε αυτή την ψηφιακή εποχή και να δείξουμε με το παράδειγμα τι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ κυρία Γιούτο. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για μια εξαιρετική πρόταση. Έχει υπάρξει μια σωστή συνεργασία για την έκθεση αυτή της κυρίας Ράνκε, γιατί περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για την πολιτική μου κίνηση, όπως η συμμετοχή των γυναικών οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, η έννοια του ε, δωρεάν διαδικτύου κτλ. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται πώς κάποιες ομάδες ε, όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε αυτές τις έννοιες τις οποίες προανέφερα έχουν ζητήσει να υπάρξει κατά ψηφούς. Λοιπόν, ε, τι τους ενοχλεί σε σχέση με τα θέματα της άμεσης δημοκρατίας στο διαδίκτυο σαν παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτή την οποία βιώνουμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε στις νέες τεχνολογίες την βοήθεια που πρέπει προς τις γυναίκες. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για διάκριση βάρος των γυναικών στην, στον ψηφιακό τομέα. Γιατί υπάρχουν ούτως ή άλλως διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και στη δύναμη, οπότε δεν νομίζω ότι ε, θα βελτιώσει και πολύ την κατάσταση των γυναικών η είσοδο στην ψηφιακή εποχή. Η κυρία Τόγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πολύ πιο σοβαρή από τον προλαλήσαντα. θα γνωρίσω πλήρως ε, τα άστοχα και ανίκια σχόλια του προλαλήσαντος. Εγώ θα μιλήσω για κάτι πιο σοβαρό, για το γεγονός ότι δυστυχώς έχουμε ελάχιστες γυναίκες στον τομέα πληροφορίας και επικοινωνίας. Και παρά τα, την πρόοδο, ακόμη έχουμε πολλές γυναίκες άνεργες στον τομέα αυτό των Επικοινωνιών και της Πληροφορίας, παρόλο που κανονικά θα έπρεπε να δίνει πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να προσλαμβάνουν γυναίκες και στον τομέα πληροφορίας και επικοινωνίας. Βέβαια, οι έξυπνοι επιχειρηματίε και εργοδότε καταλαβαίνουν την ανάγκη να διασφαλίσουν ισορροπία μεταξύ άνδρων και γυναικών, όχι μόνο για να βοηθήσουν τον κόσμο να αμείβεται για τη δουλειά του, αλλά για να βελτιώσουν την κατάσταση επιχείρησης. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη απασχόληση στις, ε, στον τομέα αυτό θα εξασφαλίσει ισότητα μεγαλύτερη μεταξύ των δύο φύλων. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μπόρεσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνει μια τόσο καλή πρόταση και θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαπερνούν κάθε ε, τμήμα της ζωής μας σήμερα και με πολύ σημαντικό μάλιστα τρόπο. Ταυτόχρονα οι ανισότητες σε επίπεδο φύλων διαπερνούν επίσης τον ψηφιακό κόσμο, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία μας παρέχει ο ψηφιακός κόσμος για να προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε τις διακρίσεις και να βοηθήσουμε τις γυναίκες ε, να γίνουν ε, ε, μεγαλύτερο κομμάτι και πιο σημαντικό κομμάτι του ψηφιακού κόσμου. Πρέπει να χτίσουμε γέφυρες επίσης ανάμεσα στην δημιουργική πλευρά από τη μία με την τεχνική από την άλλη. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την δημιουργία με την τεχνική επάρκεια. Gracias. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θετική αυτή η έκθεση και αυτή η συζήτηση και πραγματικά θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε η συγκήτρια. Πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ έχω εργαστεί στον τομέα της πληροφορικής, ανησυχώ για το πώς λίγες γυναίκες δουλεύουν ε, πραγματικά, όχι θέσεις διοικητικής υποστήριξης σε αυτό τον κλάδο. Και πρέπει να το δούμε αυτό νωρίς, στα σχολεία, στα δημοτικά, να ασχοληθούν τα κορίτσια με τα μαθήματα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να γίνουν ε, προγραμματιστές, αναλυτές κτλ. Δεύτερον, τις προάλλες μιλούσα με κάποιες ε, γυναίκες επιχειρηματίες ε, στον ψηφιακό τομέα που έφυγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήγαν στη ΣΥΠΑ. Γιατί εκεί είναι οι ευκαιρίες. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το ταλέντο των ανθρώπων αυτών. Πρέπει οι γυναίκες επιχειρηματίες ε, να είναι κάτι το οποίο παίρνουμε εξίσου σοβαρά με τους άνδρες. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε. κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε την ε, κατάσταση όσον αφορά την ισότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αξίζει να μέρει την προσοχή μας. Το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον κλάδο της πληροφορικής είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η έκθεση της κυρίας Ρέιτκε συνεισφέρει στο να αναδείξει το θέμα και έχει κάποιες πολύ καλές συστάσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον κλάδο και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο να κλείσει το χάσμα των δύο φίλων στον κλάδο αυτόν και θα ήθελα άρα να την ευχαριστήσω για την εξαιρετική αυτή έκθεση. η Κομισιόν σκοπεύει να λάβει περαιτέρω δράση όπως εξάλλου αναφέρει και η στρατηγική για την ισότητα των φίλων. Εξάλλου μεγάλος συνασπισμός ε, για το θέμα αυτό ακριβώς αντιμετωπίζει την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Κάποια από αυτά μάλιστα τα οποία έχουμε ως δεσμεύσεις αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες και ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μεγάλο συνασπισμό για να στηρίξουμε μέτρα τα οποία θα ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες ε, ε, στις γυναίκες και τα κορίτσια και βεβαίως την απασχόλησή τους στον κλάδο. Η Κομισιόν προωθεί επίσης ε, τις γυναίκες. Όπως είπαμε, ο κλάδος αυτός αυξάνεται διαρκώς, δημιουργεί 120 νέες θέσεις κάθε χρόνο. Δεδομένων των καλών εργασιακών προοπτικών θα θέλαμε να δούμε και περισσότερες γυναίκες να εκμεταλλεύονται την ε, κατάσταση αυτή και να σκεφτούν μια σταδιοδρομία στον κλάδο αυτόν. Καθώς ε, υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το ωράριο και έτσι οι γυναίκες ε, θα έχουν και μικρότερο πρόβλημα ανεργίας. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα οικονομικά επιχειρήματα, αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, η μελέτη της ε, Κομισιόν ε, όσον αφορά τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται είδε πως ε, οι γυναίκες στον κλάδο αυτών δημιουργούν κάθε χρόνο 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίζουν 9% παραπάνω από γυναίκες σε συγκρίσιμες θέσεις ε, στους υπόλοιπους κλάδους των υπηρεσιών. Για να αυξηθούν λοιπόν οι ευκαιρίες στην ψηφιακή εποχή πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υποεκπροσώπηση των γυναικών αυτή τη στιγμή. Μόνο 9 στους 100 ε, app developers ε, είναι γυναίκες στην Ευρώπη και λιγότερο από 30% του κλάδου της πληροφορικής είναι γυναίκες συνολικά. Αν δούμε λοιπόν επίσης την πλευρά της εκπαίδευσης βλέπουμε πως μόλις 29 στις ε, χίλιες γυναίκες πτυχιούχους έχουν ένα πτυχίο που έχει σχέση με τους υπολογιστές. Η Κομισιόν ε, υποστηρίζει τις ε, πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να αυξήσουν τις γυναίκες σε αυτές τις δουλειές και τις σπουδέ. Παραδείγματος χάρη. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών του Διαδικτύου είναι το πρώτο δίκτυο που στηρίζει ειδικά τις γυναίκες για να αναπτύξουν τις διαδικτυακές τους επιχειρήσεις, δημιουργεί δεσμούς μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών και προωθεί το όλο σύστημα επιχειρηματικότητας στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή ενιαία αγορά με την διάσταση της ε, ηλεκτρονικής κοινωνίας είναι μια ευκαιρία για τις γυναίκες αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα πρότυπα και ε, γυναίκες οι οποίες θα βοηθούν νέες άλλες γυναίκες να μπουν στον κλάδο και βέβαια πιο στοχευμένα προγράμματα για ε, σπουδές και εργασία στον κλάδο. Επίσης ε, περισσότερες πρωτοβουλίες όπως η εβδομάδα γραφής ε, κώδικα όπου είχαμε 500.000 νέους προγραμματιστές και κορίτσια βεβαίως μεταξύ αυτών. Και πρέπει λοιπόν να δούμε όπως είπαμε και το θέμα της πυκλομορφίας. Θεωρώ λοιπόν πως το να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα για τα φύλλα θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες και να προσελκύσουμε περισσότερες γυναίκες στον κλάδο. Όπως επίσης τονίζει η έκθεση, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση της κοινωνίας σημαίνει και κάποιες απειλές για την ισότητα μεταξύ των οποίων τον ...κύβερνο παρενόχληση... και σεξισμό. Βλέπουμε λοιπόν πως ε, Σύμφωνα με έρευνες, μία στις 10 γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή παρακολούθηση μέσω των νέων τεχνολογιών. Όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών και στο διαδίκτυο βασίζονται στις ανισότητες αυτές και τις ενισχύουν περαιτέρω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να καταπολεμήσει το πρόβλημα αυτό με κάποια στρατηγικά έγγραφα. Μια δράση που έχει αναλάβει η Κομισιόν στον τομέα αυτών είναι οι προτάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας που περιέχει διατάξεις για να ενθαρρύνει την συμμετοχή ε, των γυναικών στον κλάδο της πληροφορικής στην καταπολέμηση του φαινομένου. Μάλιστα, δεδομένων των εξαιρετικών προτάσεων που υπάρχουν σε αυτή την έκθεση, είναι σαφές ότι έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Θα πρέπει λοιπόν να εξευνήσουμε τρόπους για να προωθήσουμε την ενδυνάμωση των γυναικών. Αναμένω λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις προκλήσεις ε, για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπα, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να προωθήσουμε την ισότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση.